Ξέρετε την πληροφόρηση υπάρχει και στο δελτίο μας. Έχουμε web streaming και διερμηνία σε ορισμένες γλώσσες. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Οπότε αρχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Οπότε, ακρόαση του υποψηφίου για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για τη Γερμανία, που το ξέρουμε πολύ καλά, είναι ο συνάδελφος ε, Κλάους Χάινα Λέινε. Αν θυμάμαι καλά, συνήθως η εισηγήτρια, η κυρία Γιάλα Σέντερ, εάν το επιθυμεί μπορεί να πει δυο λόγια και μετά και μετά α όχι καλύτερα να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Λένε αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι μου δώσατε πέντε λεπτά για να επιχειρήσω να εξηγήσω γιατί θα προσπαθήσω να περιοριστώ με τρία θέματα θα ασχοληθώ με τρία θέματα γιατί λοιπόν θέλω εγώ και γιατί υπάρχει πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης να γίνω ε, μέλος του ηλεκτρικού συνεδρίου. Δεύτερον, ε, γιατί είμαι κατάλληλος και τρίτον ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς ανεξάρτητος. Είμαι 22 χρόνια ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν μου τηλεφώνησαν το Βερολίνο μετά από 22 χρόνια και μου πρότειναν να είμαι υποψήφιο τη γερμανική κυβέρνηση για αυτό το αξίωμα, δεν το σκέφτηκα πολύ. Είμαι 55 περίπου. Λογικό είναι να αποφασίσει κανείς από την ηλικία αν πρόκειται να κάνει κάτι ακόμη. Μια νέα πρόκληση μετά από 20 χρόνια. Είναι κάτι που με συναρπάζει. Δεν το σκέφτηκα λοιπόν πολύ. Και είπα βεβαίως πριν πάρω την απόφαση αυτή, πήρα κάποια πληροφόρηση για το ελεκτικό συνέδριο και κατέληξα ότι έχει σημαντικά καθήκοντα το θεσμικό αυτό όργανο. Επίσης πρέπει να μεταρρυθμιστεί σε σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας του το οποίο θα πρέπει να θέτει την ε, εργασία του στη διάθεση αυτών για τους οποίους εργάζεται. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορώ να συμβάλλω ούτω ώστε η πληροφόρηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμικών οργάνων και ιδίως μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Συνεδρίου, Ελεκτικού Συνεδρίου ε, να είναι καλύτερη και ιδίως ε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να πληροφορείται καλύτερα. Υπάρχουν ε, πολλά ενδιαφέροντα κείμενα τα οποία εκπονήσαμε για την εξέλιξη του ελεκτικού συνεδρίου. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά και ε, στα εσωτερικά έγγραφα του ελεκτικού συνεδρίου να περιλαμβάνονται. Πρέπει λοιπόν να γίνει πιο αποτελεσματικό, να αναπτυχθεί περαιτέρω το συνέδριο και εάν εκλεγώ για τα επόμενα 6 χρόνια μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα δώσω βάρος σε αυτό. Πόσο είμαι ε, κατάλληλος. Δεν ε, έχω πτυχίο οικονομικών, αλλά αυτό για τους οικονομικούς οργανισμούς ε, είναι συνηθισμένο πολλές φορές ε, ε, εργάζονται νομικοί σε αυτόν τον ε, τομέα. Είμαι και εγώ νομικός, έχω δύο νομικά πτυχία, έχω εκπαιδευτεί και ως δικαστής. Ασχολούμαι πολύ με τα δημοσιονομικά. Έχω πείρα και σε αυτά. Αυτά μπορείτε να τα εξαγάγετε και από τις απαντήσεις που έδωσα στις γραπτές σας ερωτήσεις. Η συγκεκριμένη πολιτική μου δραστηριότητα ασχολήθηκε πολύ με τα χρηματοδοτικά και δημοσιονομικά θέματα και όταν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μιας μεγάλης πόλης του Ντίσσελντορφ και όταν ήμουν μέλος της ε, Γερμανικής Βουλής ασχολήθηκα και εκεί με θέματα προϋπολογισμού και ως μέλος ε, της Επιτροπής Έρευνας για το πώς ε, εργάστηκε η Επιτροπή Ιδιωτικοποίησεων της Ανατολικής Γερμανίας και σε άλλα καθήκοντα. Εδώ τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα περιορισμένα με τα δημοσιονομικά όσο ήμουν μέλος της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Υπεροπολογισμού. Έχω ασχοληθεί όμως πολύ με λογιστικά θέματα τα τελευταία λοιπόν 20 χρόνια. Έχουμε ασχοληθεί με πολλά τέτοια θέματα και έχω υπάρξει εισηγητής για πολλά τέτοια θέματα όλες τις οδηγίες για τα λογιστικά πρότυπα λοιπόν ήμουν ε, εισηγητής για αυτές, ε, ιδιαίτερα για τα θέματα ιδιωτικού δικαίου και πέρυσι όταν αναθεωρήσαμε την τέταρτη και έβδομη οδηγία για τα θέματα που αφορούν το εργατικό δίκαιο και τα λογιστικά του. Κατά πόσον είμαι ανεξάρτητος από ό,τι ξέρω, είναι σαφείς οι διατάξεις γι' αυτό και θα τις ε, ακολουθήσω γιατί πιστεύω ότι είναι και σωστές. Όλες οι άλλες δραστηριότητες μου θα σταματήσουν. Ήδη από την επόμενη εβδομάδα θα παρεντηθώ από την θέση του Προέδρου της ε, ε, οργάνωσης ε, της, ε, του κόμματός μου στο Ντίσσελντορφ και επειδή την 1η Μαρτίου θα αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα θα ε, παρετηθώ και από όλες μου τις ιδιωτικές δραστηριότητες. Δεν θα έχω λοιπόν καμία συμμετοχή. Θα κλείσουν τέτοιες δραστηριότητες. Όπως σας είπα διευκρίνησα ότι και για, το, για τη συμμετοχή μου σε ένα δικηγορικό γραφείο όσο θα είμαι μέλος του ελεκτικού συνεδρίου δεν θα ε, έχω καμία δραστηριότητα ως δικηγόρος. Όλες τις υπόλοιπες ε, δραστηριότητες μου είτε είμαι μέλος ε, ελεκτικού, ε, συγγνώμη, εποπτικού συμβουλίου ή οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες θα τις εγκαταλείψω, θα παρατηθώ. Εάν εκλεγώ στο ελεκτικό συνέδριο θα ενημερώσω όλους τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχω ότι θα παρετηθώ. Όλες λοιπόν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία για να είναι μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και για να εργάζεται κανείς στο συνέδριο θα τις εκπληρώσω. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά και βεβαίως στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λένε. Να ακούσουμε τώρα λοιπόν την εισηγήτρια και μετά θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Καταρχήν καλωσορίζω τον κύριο Λένε στην Επιτροπή μας. Είναι γεγονός ότι είχαμε επαφές και στο παρελθόν, γι' αυτό λοιπόν θα ε, ήταν ενδιαφέρον εάν ε, τελικά εκλεγεί στο ελληνικό συνέδριο. Ε, πω το ότι έχει κάποια έλλειψη εμπειρίας σε ορισμένα στήματα. Θα ήθελα λοιπόν για το λόγο αυτό να μπορέσετε σε σχέση με όλα όσα, όσα είπατε για την πολιτική σας σταδιοδρομία να μας αναφέρετε με ποιο τρόπο διότι ανοίγω παρένθεση οι απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις που έβαλε η Επιτροπή μας κάνατε κάποιες αναφορές πολύ σωστά εξάλλου για κάποια σημεία τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον π.χ. η εμπειρία σας σχετικά με την το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας και με ποιο τρόπο πιστεύετε πως θα μπορούσατε να βοηθήσατε να βοηθήσετε το ελεγκτικό συνέδριο με βάση την εμπειρία της. Το θέμα της ανεξαρτησίας. Ε, υπάρχει θέμα σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Ε, Μείνετε πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο κατά διάρκεια της πολιτικής αδειοδομίας και ήσασταν επαΐων σε θέματα διαφάνειας. Γεγονός από το 2003 είναι πως ανήκετε σε ένα σημαντικό όργανο, δικηγορικό γραφείο και είσαστε εξειδικευμένος σε θέματα αυτής της φύσης και φυσικά η... Ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το... το βουλευτικό σας αξίωμα είχε κάποια διαφορά, σε κάποια σύγκρουση με τα επαγγελματικό σας έργο τώρα. Το θέμα είναι η σχέση που είχατε με την αναθεώρηση που έγινε για το ζήτημα του καπνού και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και δεδομένου ότι εσείς ήσασταν πρόεδρος ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ήσασταν και εισηγητής για την γνωμοδότηση σχετικά με τον καπνό. Και αυτό οδήγησε σε κάποιες αντιδράσεις, διότι το γραφείο στο οποίο ε, δουλεύατε ως ε, δικηγόρος έχει ως πελάτες μια διεθνή εταιρεία καπνού. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με ποιο τρόπο αυτή η κατάσταση θα διορθωθεί και δεν θα υπάρξει καμία σκιά που προκειμένου να επηρεάσει το έργο σας ε, ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης υπάρχει και μια σειρά άλλων ζητημάτων ειδικά με τη δραστηριότητά σας. Αναφέρεται πως ε, θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο θεσμικό σας όργανο και το Κοινοβούλιο αλλά και ειδικά με την Επιτροπή Προπολογισμού, ε, Ελέγχου Προπολογισμού της, ε, του Κοινοβουλίου αλλά θα πρέπει φυσικά όπως καταλαβαίνετε να υπάρξει μια ισορροπία έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει μια αγαστή συνεργασία. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω, τις ιδέες σας δηλαδή, γιατί σε κάποιο σημείο αναφέρεται ότι δεν ε, θα Θα ήθελα να σταματήσω στο σημείο αυτό. Τώρα, αν ο Πρόεδρος ε, μου δώσει μια δεύτερη δυνατότητα μετά από τις ε, ερωταποκρίσεις ε, των συναδέλφων και φυσικά θα ήθελα όλες αυτές οι ερωτήσεις να απαντηθούν τόσο από όσο και από τους ενδεχόμενους μεταδικούς υποψηφίους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν ε, ένα πακέτο ε, το, ε, αυτά που θέσατε ως ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω. Να ξεκινήσω με το γενικό σας ερώτημα. Το ελεκτικό συνέδριο δικαίως αποτελεί ένα θεσμικό όργανο από τους προπάτορες των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Αποτελείται από μέλη που έχουν τελείως διαφορετικές εμπειρίες, ε, υπάρχουν ε, ελεγκτές με την κλασική έννοια, υπάρχουν ε, αυτοί που έχουν συγκεκριμένες δραστηριότητε και εμπειρία σε ό,τι αφορά τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πρακτική εμπειρία από τα θεσμικά όργανα και με βάση αυτή τους την εμπειρία μπορούν να κρίνουν το πώς λειτουργούν τα θεσμικό όργανα και πού υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η συλλογική δραστηριότητα και διαχείριση του ελεκτικού συνεδρίου. Εγώ είπα από την αρχή ότι δεν είμαι το τυπικό παράδειγμα ενός ελεγκτού, ορκωτού λογιστού α πούμε, αλλά έχω την εθνική μου εμπειρία σε αυτή σας παραπέμπω, από τους 17 προέδρους, των, ε, από τους 17 ε, προέδρους του Ελεκτικού Συνεδρίου της Γερμανίας δεν είναι κανένας οικονομολόγος. 15 μάλιστα ήταν νομικοί, όπως εγώ. Και οι υπόλοιποι είχαν πολιτικό παρελθόν. Από τους 17 αντιπροέδρους των Ελεκτικών Συνεδρίων στη Γερμανία, οι 13 πάλι είναι νομικοί. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον στα μεγάλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ευρύτερη εμπειρία, ευρύτερες γνώσεις και νομίζω ότι και εγώ με την ευρεία μου εμπειρία, μιλήσατε και για, την, ε, για το ξέπλυμα ε, χρήματος, ε, μπορώ να συμβάλλω στην δουλειά αυτού του θεσμικού οργάνου. Αν δεν πίστευα ότι δεν μπορούσα να το κάνω, δεν θα είχα υποβάλει υποψηφιότητα. Τώρα, για τις υπηρεσίες και τον ρόλο που θα πρέπει να, τον, τη σχέση που θα πρέπει να έχει το ελεγκτικό συνέδριο και το, με το κοινοβούλιο. Το είχα θεωρήσει και εγώ αυτό σημαντικό σημείο. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι ο σκοπός. Έχει πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα. Αυτά τα συγκεκριμένα λοιπόν καθήκοντα, μεταξύ άλλων, είναι τα θεσμικά όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για τον προπολογισμό και για θέματα τέτοια να τα, να τα υποστηρίζει. Το Κοινοβούλιο βεβαίως είναι αυτό, έχει αυτό ως καθήκον κάθε χρόνο και γι' αυτό προετοιμάζεται από την, από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού όλη η διαδικασία για την απαλλαγή και δίδεται. Βεβαίω και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και σε ένα πλαίσιο και η Κομισιόν παρεμβαίνει ε, έτσι ώστε να μπορούν να, να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Βεβαίως το θέμα της ανεξαρτησίας είναι σημαντικό. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο είναι αυτό που τελειώνει, που αποφασίζει συγγνώμη, στο τέλος και ο βασικός του ομόλογος ε, θα πρέπει να έχει θετική αντίδραση, απάντηση. Αυτό που θέλουμε είναι η εντατικοποίηση και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε σε μια νομοθετική φάση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν ασχολούμαστε με νέα πράγματα, ασχολούμαστε κυρίως με βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Οπότε ε, θα μπορούσαν ε, τα αποτελέσματα κάποιων ειδικών εκθέσεων να βοηθήσουν πάρα πολύ τον νομοθέτη όταν πρόκειται να κάνει ε, μεταρρύθμιση της νομοθεσίας. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ε, ασχοληθούμε πολύ περισσότερο. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά σημεία. Μιλήσατε για το θέμα των δικηγορικών μου καθηκόντων. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Βεβαίω δεν είναι η παράπλευρη ασχολία μου η δικηγορική, είναι η βασική μου ασχολία. Και ξέρετε ότι οι δικέ μου παρεμβάσει σε, σε αυτόν τον οίκο πάντα βρίσκονταν, βρισκόμουν μέσα στους δύο ή τρεις πρώτους ε, υποβάλλοντες νομοδοτήσεις. Είμαι λοιπόν από τους καλούς μαθητές αυτού του οίκου. Δεν είναι λοιπόν δευτερεύουσα η δραστηριότητά μου, είναι η πρωτεύουσα αυτή αλλά ε, και ως βουλευτής ε, πάντα ήταν σημαντικό για μένα να είμαι ανεξάρτητο. Ποτέ δεν βρέθηκα ή δεν ήθελα να βρεθώ σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούσα, θα έπρεπε μάλλον να εξαρτήσω την επανεκλογή μου από το, από το κόμμα μου. Έχω βεβαίως ε, πάντα τις επαφές μου και κανείς δεν ξέρει βεβαίως τι συμβαίνει στην πολιτική. Διατηρούσα λοιπόν τις δραστηριότητε αυτές. Αν λοιπόν πρέπει να κερδίσω το ψωμί μου ως, ε, ως ε, δικηγόρο στην χώρα μου, αυτό θα, θα κάνω. Ε, η ανεξαρτησία μου όμως πάντα ήταν σημαντική για μένα. Ένα σημαντικό κομμάτι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων μου έχουν να κάνουν με, τις, ε, με το διαδίκτυο που έχω δημιουργήσει στην, στη, στη χώρα μου, στην πόλη μου. Ήμουνα δέκα χρόνια μέλος του κόμματος που διοικεί την ε, περιφέρεια αυτή. Και αυτό νομίζω ότι εξηγεί και τις υπόλοιπες δραστηριότητές μου. Για την οδηγία τώρα για το καπνό. Πριν την ψηφοφορία για την έκθεση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, εκείνο το απόγευμα, μια μη κυβερνητική οργάνωση, δεν θυμάμαι και ποια είναι, ε, έκανε στο, ε, έδωσε στο, στο ε, διαδικτύο συγγνώμη, κάποιες κατηγορίες ότι υπάρχουν, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων γιατί η δική μου η δικηγορική εταιρεία, αυτή που δουλεύω, ήταν, είχε ως πελάτη μια μεγάλη εταιρεία καπνού. Την ημέρα λοιπόν της ψηφοφορίας έγινε η ψηφοφορία, ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση, ήταν ε, πολύ ισορροπημένη, 17 προς 4 ήταν η ψήφη, αλλά ταυτόχρονα μιλήσαμε και για τους νομικούς κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε ότι μια οδηγία για τις, ε, για τις διαφημίσεις για τον καπνό έχει φτάσει μέχρι το δικαστήριο. Οπότε στο Ντουμπάι η δικηγορική μου βρέθηκε ε, ε, για την, ε, σε μια τέτοια, σε, βρέθηκε σε μια θέση να πρέπει να ε, υπερασπιστεί μια μεγάλη εταιρεία καπνού μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Η Teller είναι ε, μια δικηγορική εταιρεία που έχει 23 δικηγορικά γραφεία παγκοσμίω. Εγώ προφανώς και κανένας άλλος δεν είναι σε θέση να ελέγξει αν κάποιος από αυτούς τους ε, ε, υπαλλήλους ή κάποιο από αυτό το γραφείο έχει αναλάβει σε κάποια στιγμή κάποια εταιρεία καπνού σε κάποια χώρα. Δεν βλέπω λοιπόν καμία σχέση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων μου του γραφείου ας πούμε στο Ντουμπάι της ε, εταιρεία μας και με τις δικές μου δραστηριότητε ε, εδώ σε σχέση με την οδηγία πάντα για τον, καπνέ, για τον καπνό. Εγώ είμαι εταίρος αυτού του ε, γραφείου, είμαι εταίρος στην Γερμανική Ένωση και δεν έχω καμία σχέση με, το, τα όσα γίνονται στην, στο γραφείο στο Ντουμπάι. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εκεί. Χαίρομαι που μου θέσατε το ερώτημα αυτό για να μπορέσω έτσι και να το ξεκαθαρίσω. Επίσης, ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να πω ότι αν, είχα, αν ήξερα από πριν, σίγουρα θα είχα ζητήσει από την εκπρόσωπό μου στην Επιτροπή Νομικών ή από, την, από κάποιον άλλο συνάδελφο να κάνει την έκθεση αυτή. Αλλά βεβαίως είναι τελείως αβάσιμες αυτές οι κατηγορίες. Και βεβαίω από την έκθεση μπορείτε να δείτε τι δικέ μου γνώσει για το καπνό και ποιε ήταν οι θέσει μου στην έκθεση αλλά και στην Ολομέλεια. Και βεβαίως ε, αυτό που κάνουμε εδώ ως ε, νομοθέτες ε, πρέπει να είναι νομικό. Δεν μπορεί να, πρέπει να είναι νομικά στεγανό, δεν μπορεί να αμφισβητείτε. Αυτά μπορώ να σας πω. Πώς θα το κρίνετε βεβαίως εσείς είναι δικό σας θέμα. Αυτές οι κατηγορίες έφτασαν μέχρι τον πρόεδρο του οίκου και μάλιστα ο συνάδελφος Χέφνερ είναι αυτός που ε, είναι ο πρόεδρο αυτή τη επιτροπή ε, που ασχολείται με την σύγκρουση συμφερόντων ή με τα οικονομικά συμφέροντα. Του τα εξηγήσαμε και ξεκαθαρίστηκε η υπόθεση. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει το λόγο Ρέστορ Λοκάλιν και Μπέρεντ. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να ε, πάρουν το λόγο με αυτή τη σειρά. Είναι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που ο Σκιώδη Ζαν Πιερωτή από την ομάδα μας ε, δεν μπόρεσε να έρθει ακόμη στη Γαλλία, αλλά μου είπε να πω ότι είμαστε υπέρ της υποψηφιότητας και δεν έχουμε καμία αμφιβολία μετά τη μελέτη της υποψηφιότητας. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Το ελεκτικό συνέδριο ασχολείται με το κατά πόσον είναι νομότυπα τα νομοθετήματά μας και καταλήγει και σε ένα ποσοστό λαθών. Πολλές φορές κάνουμε λοιπόν ε, ε, συζητήσεις για τα λάθη αυτά που έχουν γίνει, τι ποσοστό έχουν και συζητάμε για κόμματα και τελείες. Είναι πολλή δουλειά. Αν θα είχαμε μία επιθυμία θα θέλαμε να περάσουμε σε πιο ουσιαστικά θέματα. Πώς είναι αποδοτική η εργασία μας. Ελπίζω με την πείρα σας από τα οικονομικά θέματα να συμβάλλετε στην εργασία του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Και η ερώτηση. Τι δυνατότητα βλέπετε να βοηθήσετε να ε, ενεργεί ταχύτερα το ελεκτικό συνέδριο. Οι ειδικέ εκθέσεις καθυστερούν πολύ. Έτσι λαμβάνουμε πληροφόρηση όταν είναι πια πολύ αργά για να αλλάξουμε την κατάσταση. Οι ειδικέ εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου με βάση τη δική μου εμπειρία την τελευταία δεκαετία ποτέ δεν οδήγησε σε ουσιώδη τροποποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί πάντα τις λαμβάναμε αργά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διευρύνει τα εργαλεία του το ελεκτικό συνέδριο και να δρά ταχύτερα. Έχει μεγάλη σημασία το ελεκτικό συνέδριο. Και πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διευρύνουμε τις δυνατότητες για να κάνουν εκθέσεις και για συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ε, λυπάμαι που χρειάζεται να το πω στους συναδέλφους. Ε, για παράδειγμα, χθε πάραμε μία έκθεση για την ε, ε, δικαιοσύνη στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα και στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι όλοι έχουν προβλήματα του ίδιου βάθους ε, που είναι το ίδιο επίγοντα. Πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε λοιπόν περαιτέρω την εργασία του ελεκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό παρακαλώ το ελεκτικό συνέδριο να μας στέλνει ταχύτερα πληροφόρηση. Ζώντε κάτι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Λένα, που ήρθατε μαζί μας σήμερα. Τρεις ερωτήσεις παρακαλώ. Πρώτη. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να εργαστείτε για το ελεκτικό συνέδριο γιατί θέλετε να αντιμετωπίσετε μια νέα πρόκληση, να αλλάξετε ε, την κατεύθυνση της καριέρας, της καριέρας σας. Καταλαβαίνω, πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη φάση της ζωής τους θέλουν μια καινούργια πρόκληση. Άκουσα επίσης να λέτε ότι αν δεν σας ε, διορίσουμε στο ελεγκτικό συνέδριο θα επανέλθετε στη δικηγορία. Δηλαδή ε, ε, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να συνεχίσετε ως Ευρωβουλευτής. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Σε δύο εβδομάδες θα εγκρίνουμε ένα ψήφισμα για το, στο, στο Στρασβούργο για το μέλλον του ελεκτικού συνεδρίου και γίνονται δηλώσεις ε, κάπως ηχηρές. Λέμε ότι τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου είναι σκόπιμο να έχουν συμμετάσχει σε εθνικά ε, συνέδρια ή έχουν ιδιαίτερη πείρα στον τομέα αυτό. Και κάπου αλλού, στην παράγραφο 4 του κειμένου μας γι' αυτό, είπαμε ότι θέλουμε υψηλού επίπεδου επαγγελματίες με πείρα στα δημοσιονομικά και ε, την ε, λογιστική των επιχειρήσεων και τον λογιστικό έλεγχο επιχειρήσεων που θα πρέπει να έχουν και πολύ καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών. Πιστεύετε ότι είναι ίσως υπερβολικά περιοριστικές αυτές οι διατυπώσεις. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε πιο ανοιχτοί ούτως ώστε να μπορούμε να διορίζουμε και άτομα με άλλο επαγγελματικό υπόβαθρο. Και τρίτη ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής συχνά εγκρίνουμε πολύ ευρείες συστάσεις. Και μετά αναρωτιέται κανείς μετά από ένα χρόνο μετά την ε, έγκρισή τους ε, τι επιπτώσεις είχαν, πώς εφαρμόστηκαν. Αν το Κοινοβούλιο λοιπόν πρόκειται να ζητήσει από το Ελεκτικό συνέδριο να περιλαμβάνει στις εκθέσεις του σε βάθος αναλύσεις των συστάσεων που έχει κάνει το Κοινοβουλίο και τι συνέχεια έχει δοθεί, αυτό θα ήταν ένα σύστημα που εσείς θα μπορούσατε να βοηθήσετε να εισαχθεί στο ελεκτικό συνέδριο εάν διοριστείτε. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ιβάηλο Κάλφιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Λένε για την παρουσίασή του. Δύο ερωτήσεις έχω να σας θέσω. Μία μπορεί να Παρεκκλίνει λίγο από αυτό που, ζήτησε, που ρώτησε ο συνάδελφος Σόντεγκρατ. ποια είναι η άποψή σας για, τις, για τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του συνεδρίου. Στο δικό σας το βιογραφικό σημείωμα Αναφέρετε ότι γνωρίζετε ποια είναι, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε τεράστια πείρα, αλλά αν δούμε Αυτά τα κριτήρια που τίθενται στην συνθήκη της Λισαβόνας είναι πολύ ευρεία. Στο μέλλον θα φροντίσετε να είναι πιο σαφή τα θέματα αυτά όπως είναι στις εθνικές πρακτικές. Ποια είναι δηλαδή τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κανείς για να γίνει μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ το ερώτημα αυτό. Δυστυχώ η απάντηση που παίρνω δεν είναι ποτέ ικανοποιητική. Για σε σχέση με τις απαντήσεις τώρα που έχετε δώσει, υποστηρίζω την πρόταση ότι στον έλεγχο συμμόρφωσης θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς συστάσει για την αλλαγή κάποιων πρακτικών ίσων ή την αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έτσι ώστε να, να μειωθούν οι δαπάνες. Πώς θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου πείτε γιατί φοβούμαι ότι με την νομική πρωτοβουλία που θα έρθει από την Κομισιόν, πώς θα μπορούσατε εσείς να, την, να κινητοποιήσετε την Κομισιόν να επιταχύνει. Ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν τον υποψήφιο. Να απαντήσω αμέσως, γιατί αλλιώς θα είναι πολλά τα ερωτήματα και ίσως να μην τα θυμάμαι έτσι λεπτομερώς όλα. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γκρέσλε. Βεβαίως είναι ένα από τα καθήκοντα του Ελεκτικού Συνεδρίου αυτό που λέτε. στα γερμανικά ελεκτικά συνέδρια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στο ιδιωτικό δίκαιο υπάρχει, αλλά στο δημόσιο δίκαιο δεν υπάρχει. Είναι θεωρητική βεβαίω η συζήτηση αυτή, γιατί υπάρχει στη συνθήκη και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η συνθήκη για αυτό. Το DAS μάλλον δημιουργεί περισσότερο παρανοήσεις Βεβαίω βοηθάει στο πώ μπορεί κανεί να κερδίσει περισσότερε γνώσει για το πώ μπορεί να βελτιώσει τι δράσει του. Εγώ προσωπικά αυτό που θα κάνω στο ελεκτικό συνέδριο είναι να υπάρξει σε πιο αυστηρό βαθμό ε, η συμπερίληψη των ε, περιφερειακών ιδιαιτερότητων. Δεν μιλάω για τι εθνικέ, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι αρκετά καυτό θέμα και στο ελεκτικό συνέδριο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο τέλο, γιατί ούτω ή άλλω έχουν συζητηθεί πολύ τα θέματα αυτά. Θα μπορούσα λοιπόν να φανταστώ ότι τουλάχιστον αν υπάρχει μεγαλύτερη συμπερίληψη των περιφερειακών ε, χαρακτηριστικών και όχι των εθνικών, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ας πούμε, κάποιες έρευνες έτσι ώστε να, γίνουν πιο λεπτο, να υπάρξουν πιο λεπτομερείς γνώσεις πάνω στο τι συμβαίνει. Η συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά ελληνικά συνέδρια βεβαίω πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα από τον, από τον ε, λογιστικό έλεγχο από τα εθνικά και τα περιφερειακά ελεκτικά συνέδρια. Πρέπει όμως να δούμε και πώς ερμηνεύονται όλες αυτές οι διατάξεις. Γενικώ πρέπει να δούμε πώς βελτιώνεται η ποιότητα. Τώρα, η κυρία Γκρέσλε μίλησε και για κάτι άλλο. Για το ότι πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι τη αποδοτικότητα. Ότι πρέπει να θέσουμε αυτό στον πυρήνα τη εργασία μα και ότι αυτό είναι και επιθυμία του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι η κατανάλωση χρόνου στο Εθνικό Συνέδριο για την ε, εκπόνηση τέτοιων ελέγχων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το είπε και η κυρία Σέντερ αυτό. Νομίζω ότι το ε, ελεκτικό συνέδριο ό,τι μπορεί να κάνει στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει πρέπει να το κάνει για να επιτευχθεί αυτή η επιτάχυνση που θέλουμε και να έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα. Για το ερωτήμα του κύριου Ζόντεγκαρτ. Βεβαίω δεν θα είμαι υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το είπα, το δήλωσα και ήδη από πέρσι και νομίζω ότι είναι σαφές από όλες τις ε, πλευρές. Τώρα, αν τα καταφέρω και περάσω, θα, θα πάω στο Λεκτικό συνέδριο. Αν δεν τα καταφέρω και δεν είμαι υποψήφιο, αν δεν με αφήσετε δηλαδή να είμαι εκεί, θα πάω στο Λουξεμβούργο τα επόμενα έξι χρόνια και θα ασχοληθώ με ό,τι ασχολιόμουν. Αλλά πάλι σα λέω ότι δεν θα είμαι υποψήφιο για τι ε, ευρωεκλογέ. Τώρα, για το θέμα των προσόντων. Διάβασα την έκθεση της κυρία Αγιάλα, ε, διάβασα και τις τροπολογίες, γιατί με ενδιαφέρουν σε ό,τι έχει να κάνει με, το, με τις μελλοντικές μου αρμοδιότητες. Αναφέρονται και οι, νομικές μου, τα νομικά μου έτσι, ταλέντα στο, κείμενο κάπου χάθηκε βέβαια, κάπου χάθηκαν κάποια από τα στοιχεία που είχα αναφέρει, στο τελευταίο κομμάτι κυρίως, γιατί η παράδοση κάποιων κρατών μελών, κυρίως αυτού που, ε, από το οποίο προέρχομαι εγώ, ε, είναι απολύτω σχετική με αυτό που θέλω να κάνω. Τώρα, αν το ε, ελεκτικό συνέδριο πρέπει να κάνει έκθεση με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Είμαι ανοιχτός ως προς αυτό. Ε, θα μπορούσα να το ζητήσω στα πλαίσια του ελεκτικού συνεδρίου, αν αυτό θεωρηθεί ότι χρειάζεται για κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Το ερώτημα τώρα του κύριου Κάλφιν, αν πρέπει να είναι πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις. Θα σου απαντήσω με μια εμπειρία μου από την, από την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Για την επιλογή των δικαστών είχαμε ένα, ε, ε, ένα φορέα για δυνάμει του άρθρου 255 της συνθήκης για να επιλεγούν. Οι ε, δεξιότητες των δικαστών βεβαίως έχουν αυξηθεί. Αυτό το βήμα ήταν πολύ πρακτικό. Αποτελείται από πρώην προέδρους ανώτατων δικαστηρίων, από εκπροσώπους των Υπουργικών Συμβουλίων και από εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου ο οποίος όμως δεν είναι βουλευτής ή μπορεί να ήταν παλαιότερα βουλευτής, αλλά έχει τις πρακτικές γνώσεις. Και αυτό σήμαινε ότι υπήρξε ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφιωτήτων και αυτό σημαίνει βελτίωση των υποψηφιωτήτων. Θα μπορούσα να σκεφτώ ότι στην επόμενη μεταρρύθμιση της συνθήκης, αυτό δεν είναι όμως θέμα να το κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, είναι θέμα των νομοθετών. Θα μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί άλλο ένα τέτοιο βήμα, γιατί πραγματικά ήταν ιδιαίτερος αποτελεσματική η δουλειά που έκανε ε, και οδήγησε σε πολύ καλή ποιοτική επιλογή των δικαστών. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να γίνει και για το μέλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό. Ε, προσπαθώ να καταλάβω και την τελευταία σας ερώτηση, την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητα της Κομισιόν. Αυτό που πρέπει να γίνει στο Ελεκτικό Συνέδριο νομίζω είναι να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος των επιτυχιών, αν δηλαδή όντως οι ε, ε, συστάσεις εφαρμόζονται αν όντω υπάρχει μετά από τις συστάσει και πράξη, αν η θεωρία γίνεται στην πράξη. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ε, εκεί θα μπορέσει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ ελεκτικού συναδρίου και κοινοβουλίου. Γιατί έτσι μπορούμε να ε, βελτιώσουμε όντως την ε, αποτελεσματικότητα και την πιο επιτυχή πολιτική. Αυτά. Ευχαριστώ. Οπότε, Τώρα έχουν ζητήσει το λόγο Ροτ Μπέρεντ και έχω βάλει και εγώ το όνομά μου. Αλλά φυσικά αν έχει κάποιος άλλος ερωτήσεις ε, θα προηγηθεί. Δεν βλέπω κανέναν άλλο συνάδελφο. Μπορείτε και αργότερα να ζητήσετε το λόγο. Η Ντάγμαρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να είμαστε ευτυχείς που έχουμε ένα υποψήφιο για το ηλεκτρικό συνέδριο που να λέγεται Καρλ Χάινα Λένε. Δεν είμαστε πάντα στη θέση να ε, επηρεάσουμε την επιλογή αυτών που ε, προτείνουν τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι κάποιος που είναι τόσα χρόνια ευρωβουλευτής που τον γνωρίζουμε όλοι όπως ε, γνωρίζουμε και τον τρόπο εργασίας του είναι καλό και χαίρομαι πολύ για την υποψηφιότητα. Πολλά ερωτήματα για την ανεξαρτησία είναι λογικό να τίθενται και ήταν σαφείς οι απαντήσεις. Όσο σαφείς μπορούσαν να είναι. Συνολικά, η ανεξαρτησία των συναδέλφων που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο και που έχουν επίσης και άλλα συμφέροντα και άλλες δραστηριότητες, ε, μπορούμε πάντα να συζητάμε πώς θα ρυθμίζεται, γιατί ξέρω πολλούς συναδέλφους που έχουν πολλές δραστηριότητες, αλλά αυτά εν παρόδο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση για το Κοινοβούλιο να εκλεγεί ο κύριος Λένε, γιατί δεν έχω και πολύ μεγάλη εκτίμηση στο ελεκτικό συνέδριο. Ίσως αυτό έχει να κάνει με το δεν είμαι τακτικό ε, μέλος της δικής επιτροπής. Εσείς όλοι μπορεί να θεωρείτε ότι είναι θαυμάσιο το ελεκτικό συνέδριο. Αλλά όταν διαβάζω τις εκθέσεις του, πολλές φορές σκέφτομαι Μα από πού έχουν κατέβει αυτά τα άτομα. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να ζει κανείς σε αυτόν τον πλανήτη με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται. Διάβασα, δεν διάβασα την έκθεση πρόοδου στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκρέσλε, αλλά διαβάζω τακτικά και πολύ προσεκτικά τις εκθέσεις ε, που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρέπει να πω ότι οι εκθέσεις αυτές καταδεικνύουν ότι οι συντάκτες τους δεν έχουν, ε, τουλάχιστον οι μισές από αυτές τις εκθέσεις, δεν έχουν ιδέα πόσο εργαζόμεθα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κάποιος ε, ε, που θα γίνει μέλος του ελεκτικού συνεδρίου να έχει πείρα ε, από το πώς δουλεύει το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς στο παρελθόν είχαμε ε, μέλη του ελεκτικού συνεδρίου ε, τα οποία είχαν διατελέσει ευρωβουλευτές αλλά ίσως δεν είχαν διατελέσει το καιρό ευρωβουλευτές ή δεν είχαν ασχοληθεί και πολύ. Ο κύριος Λένε είναι διαφορετικό και πολύ καιρό μέλος του Κοινοβουλίου είναι και πολύ ενεργό μέλος του Κοινοβουλίου. Ερώτηση τώρα. Όπως είπε ο κύριος Όντεγκαρτ και στον κύριο Κάλφιν ε, ε, και απαντώντας αυτούς είπατε ότι πρέπει να ελέγχετε πόσο έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Θέλω να πω ακόμη παραπέρα. Εάν δεν έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, δεν θα πρέπει να ελέγξει το ελεκτικό συνέδριο μήπως ήταν ανεφάρμοστες και ανόητες οι συστάσεις του. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει 50% πιθανότητα να ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε, να επανέλθω τώρα στην εργασία του Κοινοβουλίου και την έκθεσή του γι' αυτό. Η ερώτησή μου. Είστε αισιόδοξο ότι θα πείσετε τα άλλα μέλη του ηλεκτρικού συνεδρίου να καταλάβουν πώς εργαζόμαστε ότι δεν επιλέξαμε να έχουμε δύο έδρες, ότι χρειαζόμαστε διερμηνία και μεταφράσεις και πολλά άλλα τα οποία το ελεκτικό συνέδριο τα θεωρεί ε, ακριβά και όχι επαρκώς αποδοτικά. Είστε αισιόδοξο. Θα μπορέσετε να τους κάνετε να καταλάβουν τι σημαίνει να ζει κανεί σε αυτόν τον πλανήτη. Ε, δηλαδή ε, να υπάρξει μια κάποια λογική να βγουν από, το, ε, από την ε, απομόνωσή τους εκεί στο Λουξεμβούργο. Η Ανδρέας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θέσω μία ερώτηση προς τον κύριο Λέινα. Πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τις ευθύνε ε, που τις αποδίδονται βάσει των συνθήκων σε ό,τι φορά την προστασία και τον ε, έλεγχο των ε, χρημάτων των φορολογουμένων. Όταν μιλά, φτάνουμε στο ζήτημα συζητήσεων περί απαλλαγής, βλέπουμε το θέμα των παρατυπιών και των ευθύων των κρατών μέλων. Εγώ δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι πάρα πολλά προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της που τις αποδίδουν οι συνθήκες. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας πριν αυτό. Οπότε, είναι κάτι για την κυρία Ροτ θα πρέπει να υπερασπιστούμε και κάπως το λειτουργικό συνέδριο. Ο Ζάνφος λένε δεν θα αναλάβει τα καθήκοντά του με στόχο να προστατεύσουμε το κοινοβούλιο από το ελεκτικό συνέδριο. Χρειαζόμαστε το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Ροτμπέρεντ. Εφόσον ερχόσαστε κάποια φορά έστω και στα κρυφά στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολισμών θα ήταν ε, βεβαίως, ε, πολύ σκόπιμο να μιλάνε και άλλοι όπως εσείς τόσο ανοιχτά, αλλά βεβαίως έχουμε πολλές ε, ανταλλαγές απόψεων με τα μέλη του Ελεκτρικού Συνεδρίου και διαπιστώσαμε ότι είναι κανονικά άτομα που καταλαβαίνουν τις δυσχέρειες του Κοινοβουλίου. Αλλά συμφωνώ σε κάτι μαζί σας, θα ήταν πολύ καλό το ηλεκτρικό Συνέδριο να μην είναι στο Λουξεμβούργο. Όποιος είναι στο Λουξεμβούργο είναι σε ένα παράδεισο των ευλογημένων. Ίσως θα ήταν καλύτερα να είναι πιο κοντά. Λοιπόν, καλύτερα να επανέλθουμε στον υποψήφιο. Να είναι αυτό στο κέντρο των συζητήσεών μας. Η, η κυρία Ροντ Μπέρεντ επένεσε τόσο τον κύριο Λένε που του είπα ότι είναι δηλητηριασμένο το δώρο στο... του ψηθήρισα το αυτή. Αλλά κάτι ε, πρέπει να διαψεύσω ότι η κυρία Μπέρεντ ε, είναι φίλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Στο τέλος φυσικά θα ξαναδώσω το λόγο στην ε, Αγιάλα Σέντερ. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν το λόγο, να κάνω μια σοβαρή παρατήρηση και μια μίσο σοβαρή ερώτηση στον κύριο Λένε. Κοιτάξτε, και οι δύο δεν είμαστε ειδικοί για οικονομικά θέματα, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαστε και άχρηστοι. Εγώ έχω την ε, αντίληψη ότι είναι πάντα σημαντικό να είναι κανείς ε, σε θέση να εξηγήσει ε, εάν και κατά πόσον υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων στις δραστηριότητές του. Καταλαβαίνω και συμφωνώ ε, με αυτά που είπατε ότι αυτά που αναφέρθηκαν δεν μπορούν να θεωρούνται σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά επειδή χρειάστηκε να ψάξετε, ε, να βρείτε, ίσως δεν ψάχνουν όλοι να βρουν όπως πρέπει. Είπατε επίσης, αν σας κατάλαβα καλά, ότι αν δεν ε, εκλεγείτε μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου, εάν εκλεγείτε μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου, θα, δεν θα έχετε κανένα εισόδημα από ε, την ε, δικηγορική αυτή εταιρεία. Εάν εκλεγείτε, θα είστε ο τρίτος χριστιανοδημοκράτης που θα γίνει μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να σας ε, ε, ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, πόσους πρώην χριστιανοδημοκράτες ε, βουλευτές αντέχει το ελεκτικό συνέδριο. Ναι, θες κάτι να πεις τώρα ή μετά. Ωραία, αφού δεν θέλει κανένα το λόγο, η εισηγήτρια για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, αγαπητή Ντάγμαρ, νομίζω ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να αφαιρόμεθα στα άλλα θεσμικά όργανα όπως και εκείνοι ε, θέλουμε να μας φέρονται. Δεν θα ήθελα να ε, προσβάλλουμε τους άλλους. Πρέπει να φερόμεθα στους άλλους όπως θέλουμε να μας φέρονται. Και όπως είπε και ο Γιένς ήδη υπάρχουν δύο πρώην ευρωβουλευτές του ΕΛΚ που είναι μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ο κύριος Λένε θα ήταν ο τρίτος, που είναι επίσης ε, συνάδελφός μας. Και επίσης υπάρχει και ένας πρώην σοσιαλιστής ευρωβουλευτής. Οπότε θα ήταν ο τέταρτος, αν εκλεγεί ο κύριος Λένε τέσσερις πρώην ευρωβουλευτές. Είναι καλή κρίσιμη μάζα και ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια το ελεκτικό συνέδριο πολλές φορές έχει έρθει εδώ και έχει συνομιλήσει μαζί μας και έχει συνεργαστεί μαζί μας. Πολύ σύντομα να ασχοληθώ με τέσσερα θέματα. Για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων σας θυμίζω κύριε Ελένα και αυτό δεν είναι κριτική, αλλά είναι μια ευκαιρία να εξηγήσετε τη θέση σας, να σας υπενθυμίσω. Η Japan ε, Tobacco είναι η Ιαπωνική εταιρεία, αλλά δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία. Ήταν ε, στο κέντρο της προσοχής ε, των υποθέσεων που μας απασχόλησαν. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και στο μέλλον και το ελεκτικό συνέδριο. Εάν γίνεται μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, εάν το ελεκτικό συνέδριο πρόκειται να ασχοληθεί με θέματα που θα ε, ε, δημιουργούσαν σύγκρουση συμφερόντων ή θα μπορούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θέλω να σας ρωτήσω, είπατε, και έχετε απόλυτο δίκιο και το αναγνωρίζω, ότι παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, πόλη του Ντίσολντορ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο για την έκθεση του Düsseldorf και επίσης ε, ε την ασφαλιστική εταιρεία Αράκ. Ήθελα να σας ρωτήσω, αμείβεστε για αυτές τις δραστηριότητες. Ναι, γιατί συνήθως για θέματα διαφάνειας είναι σκόπιμο να μάθω αν αμείβεστε, γιατί στη δήλωση συμφερόντων σας δεν αναφέρεται. Και θέλω να τονίσω ότι μας ενδιαφέρουν πολύ οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου και είναι σημαντικό να είναι δημόσιες και να περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες για την ανεξαρτησία σας. Το είπε και ο συνάδελφος Γένς. Είστε βαρέων βαρών στέλεχος του κόμματός σας, όχι μόνο στην πόλη σας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα και εδώ στο Κοινοβούλιο και αυτό φαίνεται και από τους συναδέλφους σας που ήρθαν εδώ να σας υποστηρίξουν. Αλλά, όπως λέει η κυρία Γκρέσλε, τα μέλη του συνεδρίου θα πρέπει να μας βοηθήσουν να αποκαλύπτουμε και να ντροπιάζουμε κάποιους στο μέλλον. Αλλά ξέρετε ότι ορισμένες φορές οι μόνοι οι οποίοι καταγγέλλονται είναι οι χώρες του Νότου που αντιμετωπίζει ε, οι χώρες του Νότου που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όμως στη Γερμανία το 2012 για παράδειγμα δύο περιφερειακά προγράμματα ε, καταγγέλθηκαν και ε, ανεστάλησαν. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχει κάποια ισορροπία. Όταν σφάλουν και κάποιοι άλλοι, τουλάχιστον να αναφέρεται. Γιατί αλλιώ μας δημιουργείται η εντύπωση ότι καταγγέλλονται μόνο κάποιοι και όχι άλλοι. Και αυτό δεν είναι σωστό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, είπατε και είναι σωστό ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να έχει ανθρώπους με διαφορετική επαγγελματική πείρα. Για μένα το ότι είστε νομικός και συμφωνώ με την κυρία Ροντμπέρντ ε, είναι πολύ καλό. Αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο και τα Εθνικά Λεκτικά Συνέδρια. διότι ε, διαφαίνεται μια ε, ανάπτυξη καλής σχέσης στα εθνικά συνέδρια, ζητάνε ε, γνωμοδοτήσεις από το ελεκτικό συνέδριο για θέματα που αφορούν ευρύτερα θέματα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ρεχθεί περαιτέρω αυτή η σχέση. Θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ε, ευχαριστώ την κυρία Ροτ για τα καλά της λόγια. Καλό είναι να ακούει κανείς ε, θετικά λόγια που και που, αναμφίβολα. Το ερώτημα είναι εάν το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ε, εγώ από τις επαφές μου διαπιστώνω ότι υπάρχει ήδη αυτοκριτική και όλες οι συστάσεις που έχει κάνει το ελεκτικό συνέδριο συζητιούνται ε, με τους ε, παραλήπτες των συστάσεών του. Αλλά παρόλα αυτά, συμμερίζομαι την άποψή σας, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκεκριμένη η αντιμετώπιση. Νομίζω ότι μπορώ, μπορεί και το Κοινοβούλιο να παίξει ένα ρόλο στη συνεννόηση. Αλλά γενικότερα πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία. Δεν έχω ε, δραστηριοποιηθεί μόνο στο Düsseldorf αλλά και στο τρίγωνο Στρασβούργο, ε, Düsseldorf και Άχεν. Και έχω διαπιστώσει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η δικτύωση. Κυρία Ανδρέασεν, η Επιτροπή έχει την ευθύνη για τον προπολογισμό. Είναι σαφές τις ηθίκες. Και δεν μπορούμε να καταλήψουμε δεν μπορεί να καταλήψει η Κομισιόν αυτήν της, ε, την ευθύνη. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που έχουμε διαπιστώσει και αλλού. Ότι ένα μεγάλο τμήμα των ε, ευρωπαϊκών δαπανών, το μεγαλύτερο, δεν ε, τα διαχειρίζονται, δεν τις διαχειρίζονται οι υπηρεσίες της Κομισιόν, αλλά εθνικές και τοπικές αρχές. Και έχουμε διαπιστώσει ότι σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα, τα κυριότερα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εκταμιεύονται και χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη οι δαπάνες αυτές, τα κονδύλια αυτά. Και επαναλαμβάνω, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο σε κάποιες χώρες μέλη. Παντού υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο μία από τις προτάσεις μου θα ήταν να περάσουμε από εθνική σε περιφερειακή αντιμετώπιση για να διαπιστώσουμε πού είναι ακριβώς τα προβλήματα. Γιατί ίσως έτσι ε, να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι επισήμως αρμόδια για την εκτέλεση του προπολογισμού είναι η Κομισιόν. Τώρα για τα θέματα των εδρών της κυρίας Γκρέσλε σε πολλά κράτη-μέλη και στην Ομοσπονδική Γερμανία τα ελεκτικά συνέδρια, όπως και τα συνταγματικά δικαστήρια που στη Γερμανία το ελεκτικό συνέδριο είναι στη Βόνη και το συνταγματικό στην Καζλούι, τα ελεκτικά συνέδρια και άλλα τέτοιου τύπου σώματα είναι σε μικρότερες πόλεις για να μην είναι έτσι στη φασαρία των πρωτεύουσων και πολύ μεγάλων πόλεων. Αυτό βέβαια δεν είναι θέμα τώρα που μπορώ εγώ να το αντιμετωπίσω εγώ. Ξέρετε ότι τα θέματα των εδρών του Κοινοβουλίου είναι θέματα ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου. Αυτά τα προβλήματα βεβαίως ε, έχουν να κάνουν με την ε, συζήτηση Βρυξέλλας-Τρασβούργο. Μιλήσατε ε, για το εάν η δικηγορική μετερία Taylor έχει ένα σύστημα συμμόρφωσης. Βεβαίως έχουμε σύστημα ε, συμμόρφωσης. Δηλαδή, εάν μια εταιρεία μας ζητήσει να γίνει πελάτης μας, προσπαθούμε κάθε φορά να δούμε εάν ο πελάτης αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων με κάποιο άλλο πελάτη μας. Αλλά ξέρετε, ε, για τον καπνό, είναι σχεδόν αδύνατο να μην υπάρχει κάπου σε κάποιο άλλο τομέα της οικονομίας μια εταιρεία που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ε, έχει ε, συμφέροντα αντίθετα με μια εταιρεία καπνού. Αλλά θέλω να ξαναπώ, για να απαντήσω και στην ερώτηση της κυρίας Αγιάλα, για το ελεκτικό συνέδριο. Θα επιχειρήσω να αποφύγω ακόμη και οποιαδήποτε εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση φερόντων. Θα αποφύγω κάθε δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι κάτι αντίθετο με δραστηριότητά μου. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τη δραστηριότητα του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά και οποιονδήποτε δικαστών πρέπει να είναι κανεί πολύ πιο αυστηρό όταν είναι μέλο τέτοιων σωμάτων από ότι όταν είναι μέλο απλώ ενό κοινοβουλίου για τη δεύτερη ερώτηση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ να πω σαφώς μόλις αναλάβω τα καθήκοντά μου θα διακόψω όλες μου τις σχέσεις με το δικηγορικό γραφείο. Εκτός από τις φιλικές σχέσεις με τους συναδέλφους μου εκεί. Δεν θα έχω καμία οικονομική σχέση. Θα σταματήσω να συμμετέχω. Και αν δεν επανεκλεγώ μετά την εξαίτεια, τότε ελπίζω ότι με βάση την επαγγελματική μου πείρα θα μπορέσω να βρω κάποια άλλη δουλειά. Δεν νομίζω ότι θα έχω δυσχέρειες. Και αυτό λοιπόν πολύ εύκολα και χωρίς ε, καμία επιφύλαξη θα παρετηθώ. Το λίγο περίεργο ερώτημα τώρα, πόσα μέλη από το ΕΛΚ αντέχει το ελεκτικό συνέδριο. Τέσσερα από τα 28 μέλη είναι ευρωβουλευτές. Τέσσερα από τα 28 μέλη του ελεκτικού συνεδρίου είναι ευρωβουλευτέ. ήταν ευρωβουλευτέ. Είναι το ένα έβδομο. Νομίζω ότι είναι ακόμη ανεκτό, θα το αντέξει. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις. Βέβαια είναι λιγότεροι οι σοσιαλδημοκράτες, ίσως αυτό να έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια συγκεκριμένη στιγμή δεν υπήρχε καμία σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Τώρα όμως υπάρχουν και πάλι κάποιες, ίσως λοιπόν να οριστούν και κάποιοι σοσιαλδημοκράτε να υπάρξει περισσότερη ισορροπία μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων. Δεν έχω καμία αντίρρηση από τις αρχές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι απάντησα. Α, τώρα για την, για την αμοιβή. Αν δείτε τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, θα δείτε ότι ε, αμείβομαι για την δικηγορική μου δραστηριότητα, αλλά όχι για τις άλλες. Και αυτό έχει να κάνει με την υποχρέωση ότι όταν είναι ε, κάποιος ε, εταίρος ενός δικηγορικού γραφείου δεν μπορεί να έχει άλλες αμοιβόμενες ε, οικονομικές δραστηριότητες. Ξέρετε ότι αν έχει κανείς άλλες οικονομικές δραστηριότητες βεβαίως όλες του οι αμοιβέ θεωρούνται έσοδα του δικηγορικού γραφείου και κατανέμονται ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχή σε όλους τους εταίρους. είναι σαφές ότι ε, το μόνο ε, ε, συμβούλιο στο οποίο συμμετείχα, το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει κάποιο εισόδημα θα είναι το Συμβούλιο της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΡΑΚ, αλλά και αυτό το ποσό πηγαίνει, όπως σας είπα, στα έσοδα του δικηγορικού γραφείου. Ευχαριστώ, ελπίζω να ήμουν σαφής Ε, γιατί όλα τα δικαιωτικά γραφεία έτσι είναι οργανωμένα. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Α, η συνεργασία με τα Εθνικά Ελεκτικά Συνέδρια αναφέρθηκε βεβαίως. Νομίζω ότι όντως έχει βελτιωθεί και το βλέπετε και στις αποτιμήσεις που κάνουμε. Οι τελευταίες εκθέσεις που έγιναν για το θέμα αυτό περιέχουν πολλές προτάσεις που προέρχονται από την πείρα των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων. Πιστεύω ότι πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό είναι μια καλή παράδοση, πιστεύω ότι θα εξελιχθεί καλύτερα. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, οπωσδήποτε θα βοηθήσει να είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο γραφειοκρατική η συνεργασία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε μέλος του ελεκτικού συνεδρίου θα έπρεπε να έχει πολύ στενές σχέσεις με το εθνικό του ελεκτικό συνέδριο. Εγώ θα το κάνω. Μόλις αναλάβω θα επισκεφθώ το εθνικό ελεκτικό συνέδριο στη Γερμανία θα πάω και στα περιφερειακά ελεκτικά συνέδρια. Θα επιχειρήσω τουλάχιστον μέσα σε ένα χρόνο να τα καταφέρω για να δημιουργήσω τις επαφές που θα με επιτρέψουν να βελτιώσω τη συνεργασία και θα πρότεινα και στα άλλα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου, εάν δεν το κάνουν ήδη εδώ και καιρό, να το επιδιώξουν ούτω ώστε να υπάρχουν στενότερες επαφές βελτίωση της συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λένε. Οπότε φτάσαμε στο τέλος του σημείου αυτού, της ημερήσιας διάταξης. Τώρα θα αποφασίσουμε αμέσως, αλλά πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες μας τώρα. Οπότε θα γίνει η ψηφοφορία εδώ και κλεισμένων των θυρών και αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι παρόντες και δεν ανήκουν στην Επιτροπή ως διερμηνής, ως τεχνική, ως βοηθή, ως συνεργάτες της ομάδας, θα πρέπει να αποχωρήσουν και βεβαίως θα σας ενημερώσουμε όταν θα μπορέσετε να ξανα...